Καλημέρα, θα αρχίσουμε με τη συνεδρίαση της Επιτροπής μας. Παρακαλώ, καθίστε. Καλημέρα σε όλους. αποχές. Θα πρέπει να κάνουμε μια ηλεκτρονική επαλήθευση. Άρχεται η ψηφοφορία για την προφορική τροπολογία 3. Ψηφίζουμε ηλεκτρονικά παρακαλώ. Πέρας. Απορρίπτεται. Όχι, ζητά συγγνώμη πρόεδρος. Εγκρίνεται. 29 ε, υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Η πρώτη υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Δύο υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τρία... Όχι, προφορική τροπολογία Ένα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η τέσσερα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Και περνάμε την ε, τελική ψηφοφορία. Ηλεκτρονικά παρακαλώ, ονομαστική. Ψηφίστε παρακαλώ. Εγκρίθηκε. 17 υπέρ, μία ψήφος κατά και τέσσερις αποχές. Τώρα Στην επόμενη ψηφοφορία 61 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 61-62 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 61-63 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 61-64 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 61-65 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 61-66. Ε, στα δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 61-67. Σε δύο τμήματα. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 71-74 ε, ε, ε, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 61-77 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 61-76 σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές, Νομίζω ότι απορρίπτεται ε, έλεγχος ε, 71, 61, 76, δεύτερο τμήμα. Απορρίπτεται. Ε, 61-72, πρώτο τμήμα, όχι δεν υπάρχει. Ε, 72 υπέρ κατά αποχές ε, εγκρίνεται. Ε, 61 δεύτερο τμήμα για πρώτο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές ε, εγκρίνεται. Ε, 61 υπέρ κατά αποχές εγκρινεται 6168. 61-68 υπέρ κατά όχι, έχει καταπέσει. Γιατί εγκρίθηκε η 50. Η 51 τώρα, υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Η 69 υπέρ, το πρώτο τμήμα κατά, αποχές, εγκρίθηκε, η δεύτερο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Ε, η 69 υπέρ. Όχι, έχει καταπέσει. Ε, η 52 υπέρ κατά αποχές ε, εγκρίνεται. Η 71 υπέρ κατά αποχές ε, εγκρίνεται. 61-53 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 61-54 υπέρ κατά αποχές έλεγχος για την 6154. Σε cierra la votación. Πέρας εγκρίθηκε. Ε, η 55 ε, ε, υπέρ, κατά. Αποχές εγκρίνεται. 56 υπέρ, κατά. Αποχές εγκρίνεται. 61-57 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται 61-58 υπέρ κατά αποχές εγκρινεται 61.70 61-70 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται Τελειώσαμε με τις ψηφοφορίες Ευχαριστούμε για τη συμμετοχή σας. Ε, περνάμε στο επόμενο σημείο. Πρέπει να περιμένουμε τώρα όμως. Κάνουμε ένα διάλειμμα για το σημείο 5. Ε, η συνάντηση με την Προεδρία έχει προβλεφθεί για αργότερα και δεν έχει φτάσει ακόμη εκπρόσωπο του Συμβουλίου. Ναι, παρατέταρτο ήταν η συνάντηση. Θα κάνουμε μια, ένα διάλειμμα, πάμε να πιούμε ένα καφεδάκι και στις 10 παρατέταρτο συνεχίζουμε.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

Please, we will... We Παρακαλώ, θα ήθελα να αρχίσουμε. Καθίστε παρακαλώ. Damos comienzo con el siguiente punto del, del Συνεχίζουμε με την ε, συζήτηση του επόμενου σημείου της ημερήσιας διάταξης σε ανταλλαγή απόψεων με την ε, Προεδρία του Συμβουλίου. Ο κύριος ε, Ρίχτερ, Υπουργός Εργασίας Κοινωνικών Υποθέσεων και Οικογενειακών Υποθέσεων της Σλοβακική Δημοκρατίας, θα μας παρουσιάσει το πρόγραμμα της Προεδρίας για τους επόμενους μήνες. και έχετε τα επόμενα 15 λεπτά για την παρουσίαση και στη συνέχεια θα ακούσουμε τους εκπροσώπους των πολιτικών μονάδων, ε, συγγνώμη, ομάδων ε, κατά το όριο για δύο λεπτά έκαστος. Και θα ήθελα παρακαλώ να μην υπερβαίνετε το χρόνο σας, ε, γιατί θα θέλαμε να κάνουμε και ένα δεύτερο γύρο έρωτα-απαντήσεων. Παρακαλώ να χρησιμοποιήσετε χρηστά το χρόνο που έχετε στη διάθεσή σας. Θα ήθελα να σε ευχηθώ όμως ήδη καλή επιτυχία στην Προεδρία. Ελπίζουμε να ελοποιήσουμε και εμείς ε, σε συνεργασία με την Προεδρία τους στόχους που επιδιώκουμε υψηλότερα πρότυπα για τα ζητήματα ε, ισότητας ε, των δύο φύλων. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Καρσία Πέρες, αγαπητά μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, κυρίες και κύριοι, Πρώτα απ' όλα επιτρέψτε μου να σας ευχηθώ καλημέρα. Την 1η Ιουλίου, βεβαίως για πρώτη φορά στην ιστορία της πατρίδας μας, αναλάβαμε την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό, μια πολύ σημαντική εξέλιξη για μας, γιατί ε, όλοι θα γνωρίζουμε ότι μέχρι πριν από 20 χρόνια η Σλοβακία δεν ήταν καν παρούσα στο χάρτη της Ευρώπης. Και τώρα έχουμε την τιμή να μπορούμε να λάβουμε την ε, Προεδρία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και αυτό το πράττουμε ε, με κάθε σεβασμό και αναλαμβάνοντας πλήρως τις ευθύνες μας. Κατά τη διάρκεια της Προεδρίας θα αναζητήσουμε ε, βιώσιμες ε, επικοδομητικές λύσεις για να παρεμποδίσουμε την κατάτμιση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι δικές μας οι προσπάθειες έχουν ως στόχο το να οικοδομήσουμε και να βελτιώσουμε την εμπιστοσύνη των πολιτών προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό λοιπόν είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό για μας. Και για μένα ε, είναι μεγάλη τιμή το ότι βρίσκομαι σήμερα εδώ και το ότι μου δίνετε ευκαιρία να απευθυνθώ στην Επιτροπή σας να παρουσιάσω τις προτεραιότητές μας και τα μέτρα τα οποία προτιθέμε θα λάβουμε κατά τη διάρκεια της Προεδρίας μας. Η ανταλλαγή απόψεων, κατά την άποψή μου, είναι μια ε, θαυμάσια πρόκληση, ένα έρισμα για να επιδιώξουμε την περαιτέρω εξάλληψη ανισοτήτων ανάμεσα σε άνδρες και γυναίκες. Και θέλω να σας πω, εκτιμώ ιδιαίτερα τη δουλειά που κάνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και ιδιαίτερα η Επιτροπή σας, γιατί πραγματικά στον τομέα της ισότητας των δύο φίλων έχετε καταφέρει πάρα πολλά. Και ο δικός σας ο ρόλος ε, είναι μοναδικός. Η προτάσεις ε, και τα νομοσχέδια που καταθέτει η Επιτροπή σας ε, αποτελούν έμπνευση για τις πολιτικές που χαράσσονται στον τομέα των, που αφορά στις γυναίκες. Επίσης, καθορίζεται και τις προτεραιότητες για τη δική μας την Προεδρία. Οι και οι στόχοι της Σλοβακικής Προεδρίας στον τομέα της ισότητας των δύο φύλων και της κατάργησης των διακρίσεων, αυτά απορρέουν με κοινή δήλωση για την ισότητα των δύο φύλων. Αυτή τη δήλωση την έχουμε υπογράψει η Σλοβακία η Ολλανδία και η Μάλτα και από ε, αυτής της δηλώσεις σκοπεύουμε να δουλέψουμε ε, πολύ ε, αποτελεσματικά. Επίσης, να σας πω ότι υπάρχουν και άλλες προτεραιότητες ε, τις οποίες έχουμε καθορίσει εντάσσοντας στον τομέα της απασχόλησης και της κοινωνικής πολιτικής. Ο πρωταρχικός σκοπός ο δικός μας είναι να διασφαλίσουμε θέσεις απασχόλησης και ή δυνατόν και την ευημερία. Η δημιουργία θέσεων απασχόλησης, η γενικότερη απασχόληση αποτελούν μεγάλη προτεραιότητα για την Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και για τους πολίτες της. Και γι' αυτό το λόγο η Σλοβακική Προεδρία θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια ε, και σε επίπεδο θεσμών και σε επίπεδο κρατών μελών για να ε, εφαρμοστούν μέτρα τα οποία θα οδηγήσουν στην βελτίωση της απασχόλησης. Και εδώ θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις πλαίσιο που θα επιτρέψουν να υπάρχει μεγαλύτερη συμμετοχή των γυναικών στην αγορά. Νομίζω λοιπόν ότι όλοι σας ε, αγαπητά μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, θα συμφωνήσετε μαζί μου ότι αυτό είναι κάτι πολύ σημαντικό. Αν θέλουμε να επιτύχουμε καλύτερη ισορροπία ανάμεσα στην εργασία, ε, την οικογένεια και την ιδιωτική ζωή η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανέλαβε μια πρωτοβουλία που στοχεύει στη δημιουργία, στην ε, στο να υπάρχει μια νέα αρχή ε, όσον αφορά στη συμφιλίωση ανάμεσα στην εργασία και την οικογενειακή ζωή. Αυτό το πρόγραμμα έχει ως στόχο να ανταποκριθεί σε ε, οικογένειες με παιδιά και σε άλλα εξαρτώμενα συγγενικά μέλη έτσι ώστε να υπάρχει καλύτερη συμφιλίωση ανάμεσα στην ε, εργασία και την οικογενειακή ζωή. Και αυτό αφορά ιδιαίτερα τις γυναίκες οι οποίες διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στις ε, οικογενειακές δραστηριότητες, πολύ περισσότερο από ότι οι άνδρες. Εμείς θέλουμε να συμβάλλουμε μέσω συζητήσεων, προτιθέμεθα να οργανώσουμε και συνέδρια, θα υπάρξει ένα συνέδριο επ' αυτού του θέματος στις 20 και 21 Σεπτεμβρίου στη Μπρατισλάβα. Βασικός στόχος είναι να ανταποκριθούμε στο να υπάρχει ισορροπία ανάμεσα στην εργασία και την ιδιωτική ζωή. Ε, να υπάρχει μία ε, θετική προσέγγιση κυρίως όσον αφορά τα πρότυπα εργασίας. Ε, να λαμβάνουμε υπόψη μας και τις αλλαγές που γίνονται, ε, ψηφιοποίηση παραδείγματος χάρη. Ένας λοιπόν στόχος του συνεδρίου θα είναι να ανταποκριθούμε στην σύγχρονη τάση του να υπάρχουν επίκαιρες δυνατότητες, ευέλικτες δυνατότητες εργασίας. Να μπορεί κανείς να επιμερίζει τις ευθύνε που έχει ε, στο σπίτι του, στην οικογένειά του, με την εργασία του, να μπορεί να συμφιλειωθεί επίση επίσης οι διαφορές ανάμεσα στους άντρες και τις γυναίκες. Προσβλέπουμε στην ανταλλαγή απόψεων ε, στο να ε, αλλάξουμε, ανταλλάξουμε απόψεις για τις βέλτιστες πρακτικές ε, για τους κοινωνικούς εταίρους. Πιστεύω ότι όλα αυτά αποτελούν μια συμβολή στη συζήτηση είναι μία απάντηση στις προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε σε αυτόν τον τομέα. Δράτουμε λοιπόν τις ευκαιρίες, κυρία Πρόεδρε, αγαπητά μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, για να σας προσκαλέσω σε αυτό το συνέδριο στην Πρατισλάβα. Η άτυπη συνάντηση της Επιτροπής Κοινωνικής Προστασίας θα προηγηθεί αυτού του συνεδρίου και θα εστιάσει και αυτή η άτυπη συνάντηση στο πώς μπορεί κανείς να συμφιλιώνει και να συμβιβάζει και την οικογενειακή και την ε, ε, επαγγελματική ζωή. Θα έχουμε λοιπόν πρακτική εμπειρία, θα, έχουμε, θα ακούσουμε για τις βέλτιστες πρακτικές όσα αυτές εφαρμόζονται στα κράτη-μέλη. Επίσης, επιθυμώ να υπογραμμίσω ότι η Σλοβακική Προεδρία είναι πρόθυμη να διαπραγματευτεί ε, νέες ε, νομοθετικές και μη νομοθετικές πράξεις που αφορούν ακριβώς τη συμφιλίωση της ε, ιδιωτικής ζωής και της επαγγελματικής ζωής. Το θέμα της συμφιλίωσης, όπως σας είπα, κυρίως όταν μιλάμε για τις γυναίκες και για τις δυνατότητες πρόσβασής τους στην εργασία, αυτό το θέμα είναι πολύ σημαντικό, έτσι ώστε να υπάρχει και μεγαλύτερη οικονομική ανεξαρτησία. Έχουμε να κάνουμε με ένα σημαντικό παράγοντα, τον οποίο οφείλουμε να έχουμε κατά νου κυρίως ε, όσον αφορά στην ισότητα ανάμεσα στα δύο φύλλα. Εμείς λοιπόν προτιθέμεθα να βοηθήσουμε έτσι ώστε να επιτευχθούν οι στόχοι του 2020, δηλαδή να μειωθεί τουλάχιστον κατά 20% ο αριθμός των ανθρώπων που εκτίθενται στις απειλές της φτώχειας ε, και ε, της κατάργησης του κοινωνικού αποκλεισμού. Η κατάσταση βέβαια είναι δύσκολη, ε, πολλοί προσπάθησαν να πετύχουν το στόχο, αλλά συνέβη ακριβώ το αντίθετο. Απομακρύνθηκαν από αυτόν. Εξάλλου, καλωσορίζουμε και την έκθεση η οποία ελέγχει θέματα που έχουν σχέση με την εφαρμογή της πλατφόρμας του Πεκίνου. Εκεί γίνεται λόγος για τις γυναίκες και για την ισότητα. Και το θέμα αυτό ε, εστιάζει την προσοχή του και στο θέμα της φτώχειας, γιατί περισσότερο πρόκειται για γυναίκες και φτώχεια, όχι γυναίκες και ισότητα. Γυναίκες λοιπόν και άνδρες, οι οποίοι πλήττονται από αναπηρία, έχουν ε, διάφορα άλλα προβλήματα. Μιλάμε και για την ομάδα των Ρωμά, ε, υπάρχουν πολλά θετικά στοιχεία που προκύπτουν ε, από την έκθεση. Έχουν σχέση με την ηλικία, με την αναπηρία, με το αν είναι κανείς επιλέξιμος. Εμάς ε, μας έχουν εμπνεύσει και οι δραστηριότητες της δικής σας της Επιτροπής. Και αυτό φαίνεται και μέσα από ένα ψήφισμα που αφορά στην κατάσταση των γυναικών. Συμπελαμβάνονται και οι γυναίκες με αναπηρία, οι πρόσφυγες και επίσης οι Ρωμά. Όλα αυτά καθιστούν ένα πολιτικό πλαίσιο. Αυτοί είναι οι παράγοντες οι οποίοι επηρεάζουν ε, θέματα κοινωνικής συμμετοχής και φτώχειας. Και εμείς θα ασχοληθούμε με τα θέματα αυτά η φτώχεια σε αυτήν την έκθεση ε, ερμηνεύεται ως ε, μια ευρεία έννοια, πολυδιάστατη. Άρα δηλαδή έχουμε να κάνουμε με περιορισμένη πρόσβαση σε κοινωνικές και άλλες δραστηριότητες. Και υπάρχουν και φραγμοί που έχουν σχέση με την κοινωνική συμμετοχή και την κινητικότητα. Η λεπτομερής ανάλυση των δεδομένων ε, οδήγησε στο να υπάρχουν πολιτικές συστάσεις σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η έκθεση λοιπόν μας δίνει ε, επικαιροποιημένους δείκτες όσον αφορά τη φτώχεια για να μπορούμε να μελετήσουμε όλα αυτά τα θέματα με περισσότερες λεπτομέρειες και πάντα με βάση τη διάσταση του φύλου. Επί τη βάση λοιπόν της έκθεσης και των συστάσεων θα ε, προετοιμαστούμε για το Συμβούλιο ΕΨΟ, ε, θα προετοιμαστούμε για τις προτάσεις του Συμβουλίου όπου ε, θα εξεταστούν οι αρνητικές επιπτώσεις στη ζωή των ανδρών και των γυναικών σε διάφορες φάσεις της ζωής τους. Γίνεται λόγος για τις ευκαιρίες που τους προσφέρονται. Εμείς λοιπόν θα εστιάσουμε την προσοχή μας κυρίως σε ε, ομάδες ε, στις κοινωνίες μας που είναι μειονεκτούσες ομάδες. Μας ενδιαφέρουν βεβαίως, ε, βεβαίως ιδιαίτερα οι μειονεκτούσες γυναίκες γιατί αντιμετωπίζουν πολλές φάσεις της διακριτικής μεταχείρισης και παρά τα μέτρα που έχουν ληφθεί για να βοηθηθούν οι γυναίκες αυτές με βάση τις ε, συστάσεις εμείς επιθυμούμε να εστιάσουμε την προσοχή μας ε, ε, στα συμπεράσματα θα εστιαστούμε θα στοχεύσουμε κυρίως στις γυναίκες Ρωμά που πλήττονται κυρίως από τη φτώχεια. Θέλουμε να βελτιώσουμε την κατάσταση των νέων Ρωμά στην Πρωτισλάβα στις 10 ε, και 11 Οκτωβρίου θα λάβει η χώρα ε, μια συνάντηση υψηλού επίπεδου. Και για μένα κυρία Πρόεδρε και αγαπητά μέλη είναι μεγάλη τιμή το να μπορώ να σας προσκαλέσω σε αυτή την ε, συνάντηση υψηλού επίπεδου. Κατά τη διάρκεια της Προεδρίας μας θα συνεχίσουμε τη δουλειά προηγούμενων Προεδριών, κυρίως αναφορά τις διαπραγματεύσεις στο Συμβούλιο στον τομέα της ισότητας και της μη διακριτική μεταχείρισης. Θέλουμε να εστιάσουμε την προσοχή μας κυρίως σε δύο προτάσεις. Ευρωπαϊκή πράξη προσβασιμότητας. Αυτή είναι μια οριζόντια οδηγία και βασίζεται στην πρόταση σχετικά με την ίση μεταχείριση. Οι πρώτες συζητήσεις που αφορούν σε αυτές τις ε, νομοθετικές πράξεις έχουν ήδη λάβει χώρα τον Ιούλιο αυτού του έτους. Ο δικός μας ο στόχος της διαπραγματεύσης είναι να επιτύχουμε τη μέγιστη δυνατή πρόοδο. Και μπορώ να σας ε, διαβεβαιώσω ότι θα συνεχίσουμε ε, την προσέγγιση των διαπραγματεύσεων με απόλυτη σοβαρότητα. Θέλουμε να καταβάλουμε ιδιαίτερε προσπάθειες, κυρίως για την πράξη ε, προσβασιμότητας. Οι διαπραγματεύσεις εξακολουθούν να βρίσκονται σε ε, αρχική φάση και εμείς θα στοχεύσουμε κυρίως στα θέματα που είναι ανοιχτά, που είναι καθοριστική σημασία για τι διαπραγματεύσει, παραδείγματος χάρη πεδίο εφαρμογής της πρότασης, ε, θέματα ορισμού, ε, θέματα ε, ρητρών και εξαιρέσεων, θέματα προσβασιμότητας. Εμείς στις διαπραγματεύσεις θέλουμε να προχωρήσουμε για να βελτιωθεί και η θέση των ατόμων με αναπηρία. Μας ενδιαφέρει να ενταχθούν πλήρως τα άτομα αυτά στην κοινωνία. Εξάλλου, η πρόταση ε, πρέπει να ε, οδήγει και σε βελτίωση της ε, ίσης μεταχείρισης όσον αφορά στον τομέα της παροχής υπηρεσιών, κυρίως εκεί. Πάντα κάτω από το πρίσμα και έχοντας κατά νου τα άτομα με αναπηρία και την Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα Ατόμων με Αναπηρία. Η ομάδα υψηλού επίπεδου για την ισότητα των δύο φύλων θα συνεδριάσει στην Μπρατισλάβα στις 7 και 8 Σεπτεμβρίου και προτιθέμετα να διεξάγουμε και περαιτέρω συζητήσεις για το πώς είναι η κατάσταση στις εταιρείες οι οποίες ε, έχουν ενταχθεί στο χρηματιστήριο. Μας ενδιαφέρει η διάσταση του φύλου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Κινητήρια δύναμης για μας θα είναι η ομάδα υψηλού επίπεδου στην Πρατισλάβα, όπως είπαμε, 7 και 8 Σεπτεμβρίου. Αυτή η ομάδα υψηλού επίπεδου θα ασχοληθεί και με την έκθεση του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου για την Ισότητα των Δύο Φύλων. Ε, το θέμα με το οποίο θα ασχοληθούν είναι γυναίκες και φτώχεια. Υπάρχουν και άλλες δραστηριότητες στον τομέα ε, της εργασίας, της απασχόλησης, κοινωνικές επιπτώσεις. Υπάρχουν τα συμπεράσματα του Συμβουλίου για την πρωτοβουλία για τους νέους και αυτά ε, υποτίθεται θα βελτιώσουν την κατάσταση νέων ανδρών και νέων γυναικών. Και εμείς θέλουμε να αξιολογήσουμε και την επιτυχία ε, του προγράμματος για τους νέους, εγγύηση για τους νέους. Ε, περιμένουμε τα αποτελέσματα της συνάντησης των αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων στην Πρατισλάβα γιατί εκεί θα κριθεί και το πώς θα χρηματοδοτηθούν τα προγράμματα του μέλλοντος. Ήδη χτες στην Επιτροπή Απασχόλησης συμφωνήσαμε επί του γεγονότος ότι αυτή η βοήθεια είναι απαραίτητη. Πρέπει λοιπόν να διασφαλίσουμε ότι η βοήθεια αυτή θα προσφέρεται στους νέους στο μέλλον. Θέλουμε επίσης να ανοίξουμε και τις ε, συζητήσεις ε, που αφορούν στην μακροχρόνια ανεργία στο Συμβούλιο. Και θέλω να σας διαβεβαιώσω, να διαβεβαιώσω ότι θα συνεργαστούμε στενά με την Κομισιόν προκειμένου να εφαρμοστούν νέα μέτρα για την αντιμετώπιση των ανισοτήτων στην ε, κοινωνία. Η στρατηγική ε, δραστηριοποίηση για την ε, ισότητα των φύλων στο διάστημα 2016-2020 είναι ένα από τα βασικά έγγραφα που έχουμε στα χέρια μας για την ενίσχυση της ισότητας των φύλων τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και σε εθνικό επίπεδο. Έχουμε συμφωνήσει σε, με την κυρία, με την Επίτροπο Γιώροβα ότι για την Προεδρία της Σλοβακίας αλλά και για ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση ένα από τα βασικά ζητήματα που μας απασχολούν είναι η καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών και θα υποστηρίξουμε κάθε προσπάθεια της Κομισιόν που θα στρέφεται προς αυτόν τον στόχο. Θέλουμε επίσης να ενισχύσουμε τη συνεργασία των κρατών μελών. Θα συνεχίσουμε τις διαπραγματεύσεις που έχουν ξεκινήσει ήδη με αντικείμενο την σύμβαση ε, της, του Συμβουλίου της Ευρώπης και, της, τη σύμβαση της Κωνσταντινούπολης για τα δικαιώματα των γυναικών και την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών. Αυτά τα ζητήματα μας απασχολούν ιδιαίτερα και γι' αυτόν τον λόγο ε, αποτελούν και έναν από τους στόχους της ευρωπαϊκής ε, ε, ε, εξωτερικής δράσης. Στόχος μας είναι να εξασφαλιστούν τα ανθρώπινα δικαιώματα των γυναικών και με βάση την επίτευξη των στόχων της χιλιετίας. Πλατφόρμα του Πεκίνου και τις δεσμεύσεις που προκύπτουν από την πλατφόρμα για την εξάλληψη της ανισότητας των γυναικών. Επίσης, στην 63η συνάντηση γυναικών που θα γίνει τον Μάρτιο στη Νέα Υόρκη, θα συμμετάσχουμε εμείς ως ε, ε, Πρόεδροι για να ε, συζητήσουμε τα θέματα εργασίας των γυναικών και θα σας παρουσιάσουμε τα συμπεράσματα που, στα οποία θα καταλήξουμε. Κύριε Πρόεδρε, αγαπητά μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, θα ήθελα να εκφράσω την ελπίδα μου αλλά και την πεποίθησή μου ότι μέσω των κοινωνικών των κοινών μας προσπαθειών θα μπορέσουμε να προσεγγίσουμε τουλάχιστον λίγο περισσότερο την πραγματική ισότητα των δύο φύλων. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την προσοχή σας και ζητώ συγγνώμη αν ε, μακρηγόρησα και μίλησα περισσότερο από όσο έπρεπε. Ευχαριστούμε για την παρουσίασή σας. Ε, γύρατε διάφορα ζητήματα τα οποία μας απασχολούν και μας ε, εδώ στην Επιτροπή των Δικαιωμάτων των Γυναικών. Ελπίζουμε να υλοποιηθούν οι στόχοι που θέσατε. Δυστυχώς, με τις ε, διαδοχικές προεδρίες παρατηρούμε με, με την ίδια στοχοθεσία μεν, αλλά ε, δεν υπάρχει, δεν σημειώνεται πρόοδος. Υπάρχουν κολλήματα που μας εμποδίζουν, δεν μας αφήνουν να υλοποιήσουμε τους στόχους ε, που θέτουμε. Ας ακούσουμε, ελπίζουμε να έχετε καλύτερη τύχη. Κύριε Ζαμπόσκα από το ΕΛΚ. Ευχαριστώ πολύ που μου δίνετε το λόγο. Σας καλωσορίζω κύριε Υπουργέ στην Επιτροπή μας. Εγώ είμαι μέλος αυτής της Επιτροπής εδώ και 13 χρόνια και στην τελευταία θητεία είχα και την τιμή να προεδρεύω της Επιτροπής αυτής. Είναι πολύ ενδιαφέρον να παρακολουθείς κανείς πώς αλλάζει η θέση της ε, γυναίκας στην κοινωνία. Αναφερθήκατε σχεδόν σε όλους τους τομείς στους οποίους αναφέρθηκε και η πρόεδρος της Επιτροπής μας. Οπότε αναμένουμε να σημειωθεί μεγάλη πρόοδος στην πράξη. Γιατί οι εκθέσεις που συντάσσουμε εμείς και που επικαιροποιούμε πάντοτε επικεντρώνονται στα ίδια θέματα. Θα θέλαμε να δούμε και λύσεις. Θα ήθελα να σας θέσω δύο ερωτήσεις που αφορούν τις ίσες ευκαιρίες. Στη συνεδρίαση των Υπουργών Κοινωνικών Υποθέσεων αναφέρατε και τις δημογραφικές αλλαγές και τις επιπτώσεις που αυτές θα έχουν στα συστήματα κοινωνικής ασφάλισης. Γνωρίζουμε ότι ένας από τους λόγους της μείωσης των γεννήσεων στον έναν στον άλλον βαθμό σχετίζεται η μείωση αυτή με φαινόμενα όπου εργοδότες δεν επιθυμούν να προσλάβουν γυναίκες λόγω της πιθανότητας να αποκτήσουν παιδιά. Εσείς τι σκοπεύετε να κάνετε για να βελτιωθεί η κατάσταση των γυναικών που είναι και μητέρες και πώς θα μπορούσαμε να βελτιώσουμε την κατάστασή τους στην αγορά εργασίας. Το δεύτερο ερώτημα μου είναι σχετικό με το πρώτο ερώτημα. Η ισότητα ανδρών και ε, γυναικών ε, αποτελεί θέμα που αναφέρεται σε πολλές ε, πράξεις και συμφωνίες εδώ και 60 χρόνια. Στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος εμείς επικεντρωνόμαστε και στο συνταξιοδοτικό χάσμα μεταξύ ανδρών και γυναικών. Θεωρούμε ότι αυτό το ζήτημα είναι ύψης της σημασίας για την επίτευξη της πραγματικής ισότητας μεταξύ των δύο φύλων. Τι σκοπεύουν να κάνουν οι υπουργοί για να χειριστούν το συγκεκριμένο θέμα και τι θα κάνει η Προεδρία σας επί του θέματος αυτού. Πώς Δηλαδή θα μπορέσουμε να ξεπεράσουμε τις διαφορές μεταξύ ανδρών και γυναικών σε αυτόν τον τομέα. Αναφέρομαι πάντοτε στο χάσμα, στο μισθολογικό και το συνταξιοδοτικό. Ευχαριστώ. Θα πρέπει να μην υπερβαίνουμε το χρόνο ομιλίας ε, γιατί δεν θα ε, προλάβουμε να μιλήσουμε όλοι. οι Σοσιαλιστές. Ευχαριστώ κύριε Υπουργέ που βρίσκεστε εδώ. Παρακολούθησα με προσοχή ε, την ομιλία σας και θα ήθελα να σας υποστηρίξω σε όλα όσα είπατε. Ωστόσο, ε, ανησυχώ γιατί τα λόγια ε, της Προεδρίας δεν καταδεικνύουν καθόλου ότι η πολιτική για τις γυναίκες θα αποτελέσει προτεραιότητα τα, τους επόμενους έξι μήνες. Τα αναφέρετε αυτά τα θέματα, αλλά στην δήλωση της Προεδρίας τα ζητήματα των γυναικών και του φίλου δεν αναφέρονται καν. Ελπίζω να μην είναι εξηχαμένοι μήνες για τις γυναίκες αυτοί. Στο πλαίσιο του τρίου προεδριών θα ήθελα να σας ρωτήσω αν θέλετε να δραστηριοποιηθείτε ε, για την ε, οδηγία για τα διοικητικά συμβούλια και αν θα ε, ε, μπορέσετε να υποστηρίξετε τη δική μας πρωτοβουλία για τη ως επαγγελματικής και προσωπικής ζωής. Στο Συμβούλιο όλα τα κράτη-μέλη έχουν ε, δεσμευτεί να ε, υπάρξει και μια στρατηγική για την ισότητα των φύλων αλλά δεν έχει ακόμη ληφθεί συγκεκριμένη απόφαση επί του θέματος. Και ως εισηγήτρια θα ήθελα να υπενθυμίσω ε, για άλλη μια φορά ότι είχε υπάρξει συμφωνία στο Συμβούλιο, στο Συμβούλιο. Και θα ήθελα να σας παρακαλέσω εσείς να αναλάβετε κάθε προσπάθεια προκειμένου να αποκτήσουμε μια στρατηγική για την ισότητα. Η κυρία Χάνιμπαλ είναι επίσης εδώ, ε, οπότε θα μιλήσει εκείνη για, το ζήτημα για τα ζητήματα των προσφύγων. Αλλά θα ήθελα να μιλήσω για την σύμβαση της Κωνσταντινούπολης. Είπατε ότι θα ε, δραστηριοποιηθείτε αποτελεσματικά προκειμένου να καταπολεμηθεί η βία κατά των γυναικών. Και αποσαφηνίσατε με τα λόγια σας ότι θα δραστηριοποιηθείτε ώστε όχι το κάθε κράτος μέλος ξεχωριστά, αλλά ολόκληρη η, Ευρώπη να υπογράψει την σύμβαση της ε... Ε... Κωνσταντινούπολης και να κυρωθεί η συγκεκριμένη σύμβαση. Νομίζω ότι είναι ένα φάρο η συγκεκριμένη σύμβαση, την οποία μετά από τόσα χρόνια συζητήσεων πραγματικά τον χρειαζόμαστε. Το λόγο λοιπόν έχει κυρία Φινάντσκα. Κοιτάξτε, θα ήθελα και εγώ να σας καλωσορίσω Κύριε Υπουργέ, σας καλωσορίζω εκ μέρους του πολιτικού μου κόμματος, της πολιτικής ομάδας του ECR. Ε, και θέλω να ρωτήσω τα εξή. Άκουσα με μεγάλη μου χαρά να λέτε ότι η γυναική φτώχεια θα είναι ένα θέμα προτεραιότητας για τη Σλοβακική Προεδρία. Όλοι μας γνωρίζουμε ότι οι γυναίκες εκτίθενται περισσότερο στη φτώχεια από τους άντρες. Αυτό αφορά κυρίως τις βέστες ε, ε, ομάδες, ε, τις γυναίκες μονογονικές οικογένειες, αυτές που φροντίζουν τα ανάπηρα παιδιά τους. Να σας πω λοιπόν ότι σε εμά αυτή τη στιγμή οι γυναίκες οι τελευταίες που φροντίζουν τα παιδιά τους ανάπηρα παίρνουν 220 ευρώ. Αυτό δεν είναι κακό, αλλά θα ήθελα όμως να σας ρωτήσω, πιστεύετε ότι αυτά τα 247, 220, 247 ευρώ το μήνα είναι ένα αξιοπρεπές ποσό για να μπορούν οι γυναίκες ε, να ζουν με τα χρήματα αυτά, μα δεν είναι εκτεθειμένες στη φτώχεια. Και η δεύτερη ερώτησή μου έχει και αυτή σχέση με τη φτώχεια. Θέλω να σας ρωτήσω, πώς ακριβώς ε, προτίθεστε να αντιμετωπίσετε το πρόβλημα της φτώχειας Πώ αντιμετωπίσετε το θέμα της γυναικείας πτώχειας κυρίω. και η τελευταία μου ερώτηση έχει σχέση με τι συμφιλίε μεταξύ δουλειάς και ιδιωτική ζωής. Ε, πολύ συχνά στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο διαπιστώνουμε ότι οι γυναίκες ευρωβουλευτίνες έχουν το δικαίωμα να φέρουν τα μωρά τους στις αίθουσες συνεδριάσεων. Όμως στο Σλοβακικό Κοινοβούλιο αυτό απαγορεύεται. Και ε, χαίρομαι που μιλήσατε εσείς, στηρίξατε μία συνάδελφο στο Σλοβακικό Κοινοβούλιο που έφερε το μωρό της, ε, της το επιτρέψατε, ε, μάλλον τη στηρίξατε και είπατε ότι θα κάνετε ό,τι μπορείτε έτσι ώστε οι βουλευτίνες ε, στο Κοινοβούλιο της Σλοβακίας να μπορούν να παίρνουν τα μωρά τους στις αίθουσες συνεδριάσεων. Και επειδή τώρα είναι η φάση όπου επικαιροποιείται και ανανεώνεται λιγάκι ο κανονισμός ε, στο Σλοβακικό Κοινοβούλιο, μπορούμε να περιμένουμε ότι εσείς και το κόμμα σας θα μας στηρίξετε έτσι ώστε να γίνει πραγματικότητα τελικά αυτή η πρόταση. Ευχαριστώ. Δεν θέλω τώρα να εμπλακώ εγώ σε εθνικά ζητήματα, όμως πιστεύω ότι είναι μια καλή πρωτοβουλία. Εάν κατάλαβα καλά, ο στόχος είναι να εγκριθεί μια τροπολογία ούτως ώστε οι βουλευτίνες ε, να μπορούν να φέρνουν στο ημικύκλιο τα παιδιά τους. Και επειδή θέλουμε ε, την ισότητα των δύο φίλων, ε, καλό θα ήταν και οι άντρες να έχουν αυτή τη δυνατότητα και να μοιράζονται τις ευθύνες. Ευχαριστώ κυρία Μινέρ. Ναι, αυτό ήθελα να τονίσω, ότι έχουν και μητέρα και πατέρα τα παιδιά. Καλό θα ήταν να δούμε και κανέναν υπουργό με παιδί σε συνεδρίαση. Να μην έχουν μόνο οι γυναίκες αυτό το δικαίωμα. Θα ήθελα να τονίσω κάτι που αναφέρθηκε ήδη ε, ε, από τους φιλελεύθερους και το αναφέρατε και εσείς ότι θα επισπεύσετε τη διαδικασία κύρωσης ε, της σύμβασης της Κωνσταντινούπολης και όπως είπε και η Μαρία Νόχιλη συνάδελφος, τονίζω κι εγώ πως ε, οι φιλελεύθεροι είναι, ε, υποστηρίζουν πάρα πολύ την κύρωση της σύμβασης. Και λυπούμεθα που δεν την έχει κυρώσει η Σλοβακία ακόμη αυτή τη σύμβαση. Ποια συγκεκριμένα βήματα θα αναλάβετε για να επισπεύσετε και η Ρωσία αυτής της ε, εκτενούς ε, ε, παγκόσμιας συμφωνίας για την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών και της ενδοοικογενειακής βίας. Δεύτερον, προς μια διαφορετική κατεύθυνση. τα συμπεράσματα του Συμβουλίου για τους ΛΟΑΔΜ τέλη Ιουνίου είναι μια επιτυχία. Ε, υπάρχει μη, λοιπόν μια πολιτική συμφωνία στα 28 κράτη-μέλη για να ε, έχουμε μεγαλύτερη ευαισθητοποίηση για τα δικαιώματα των ΛΟΑΔΜΑ. Η συμφωνία του Ιουνίου ε, ισοδυναμεί με δέσμευση για αιτήσια έκθεση από πλευράς των κρατών μελών σε σχέση με την κατάσταση για τα δικαιώματα των ΛΟΑΔΜ, ούτως ώστε να δούμε που εξακολουθούν να υπάρχουν προβλήματα και να βρεθούν οι κατάλληλες λύσεις. Αυτό ελπίζουμε θα ενισχύσει τη θέση των ΛΟΑΔΜ σε ολόκληρη την Ευρώπη. Ε, τέλη του 2016 αναμένει την πρώτη έκθεση προόδου. Ποιε πρωτοβουλίε σα ρωτώ λοιπόν να λαμβάνει η Σλοβακική Προεδρία ούτω ώστε να παραμείνει ψηλά στο Ευρωπαϊκό Θεματολόγιο αυτό το ζήτημα. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Από την ΚΟΥΕ κυρία Βιόρκ. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να σας καλωσορίσω στην Επιτροπή μας, εδώ στο Κοινοβούλιο. Είπαν οι συνάδελφοι ήδη ότι θα πρέπει να καταπολεμήσουμε τη βία κατά των γυναικών και θέλουμε να σημειωθεί πρόοδος με τη σύμβαση της Κωνσταντινούπολης και φυσικά θα εμπλεκόμαστε στις προσπάθειες που γίνονται εδώ στην Επιτροπή μας. Εγώ θέλω να τονίσω το εξής. Καλά είπατε ότι θα πρέπει να εστιάσουμε και στο θέμα της ένδυας των γυναικών. Συμφωνούμε λοιπόν αυτό σχετίζεται με τις πολιτικές ε, που ακολουθούμε για την οικογενειακή ζωή και τη συμφιλίωσή της με την επαγγελματική ζωή. Χρειαζόμαστε καλύτερη νομοθεσία σε ευρωπαϊκό επίπεδο για να συνδυαστεί η οικογενειακή και επαγγελματική ζωή τόσο για τις γυναίκες όσο και για τους άντρες. Ε, ε, θα πρέπει να υπάρξει ισότιμος καταμερισμός των ε, καθηκόντων. Χρόνια τώρα συζητούμε αυτό το ζήτημα και ελπίζουμε να δώσετε μια νέα όθηση από τη διάρκεια της Προεδρίας σας. Ε, επίσης, το θέμα της περίθαλψης των παιδιών για κάποια σημεία έχει συμφωνήσει το Συμβούλιο, αλλά δεν υπάρχει επικαιροποίηση και δεν υπάρχει καμία πολιτική όθηση θα θέλαμε και πάλι να ενισχυθούν οι φιλοδοξίες σε σχέση με την ενίσχυση των συστημάτων περίθαλψης των παιδιών στην Ευρώπη. Για την ένδυα των γυναικών θα πρέπει να έχουμε το θάρρος να θέσουμε το δάκτυλο επί του τύπου των Έχουμε τις γυναίκες μετανάστριες θα πρέπει να δούμε ε, αυτές τις γυναίκες, αυτά τα κορίτσια που προσπαθούν ε, να ξεφύγουν από τον πόλεμο και από τη δίωξη να έχουν ε, πρόσβαση στις απαιτούμενες υπηρεσίες. Χρειαζόμαστε μια οικονομική πολιτική ταυτόχρονα που δεν υπονομεύει όμως τη θέση των γυναικών και των κοριτσιών στην κοινωνία. Και τέλος, αλλά εξίσου σημαντικό για την Επιτροπή μας, θα πρέπει να προωθηθεί για το ζήτημα της σεξουαλικής και αναπαραγωγικής σεξουαλικής υγείας, όχι μόνο για τις γυναίκες και τα κορίτσια, αλλά και για τους άντρες και για τα αγόρια. Θα πρέπει να έχουμε αυτοδιάθεση του σώματός μας. Αν δεν το καταφέρουμε αυτό, δεν πρόκειται ποτέ να προοδεύσουμε στην Ευρώπη. Ευχαριστώ πολύ και τώρα εκ μέρου των Πρασίνων ο κύριος Έρανστε Ούρτερσον. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε που είστε μαζί μας. Σας ευχαριστώ και για την παρουσίαση. Πολλοί από εμά έχουμε την αίσθηση ότι το ζήτημα του, της ισότητας των ε, φύλων ε, έχει ε, αντιμετωπίσει διάφορα εμπόδια και ότι δεν προχωράει το τελευταίο διάστημα. Ε, είναι σημαντικό να το γνωρίζει αυτό η Προεδρία σας και θα ήθελα να συμφωνήσω και με τις παρατηρήσεις που έκαναν άλλοι συνάδελφοι μας απογοήτευσε δηλαδή ε, σε έναν βαθμό το γεγονός ότι στο κρατό σας πρόγραμμα δεν αναφέρεται τίποτα για την ισότητα των φύλων. Παρ' όλα αυτά έχει την ευκαιρία να κάνετε πολλά πράγματα. Μπορείτε να επισπεύσετε την διαδικασία κύρωση τη Σύμβαση τη Κωνσταντινούπολη. Υπάρχουν δύο νομοθετικοί φάκελοι που μας ενδιαφέρουν και θα θέλαμε να μάθουμε αν εσείς σκοπεύετε να αναλάβετε ε, δράση προκειμένου να επιφεύσετε την, ε, ε, την διαδικασία των διαπραγματεύσεων. Υπάρχουν και το, υπάρχει και το ζήτημα των γυναικών στα διοικητικά συμβούλια. Θα θέλαμε να μάθουμε αν σκοπεύετε να κάνετε οτιδήποτε, γιατί στην Επιτροπή μας θέλουμε να προχωρήσει ο συγκεκριμένο φάκελος. Και δεύτερο θέμα, όπως γνωρίζετε, ε, μας λύπησε ε, το γεγονός της απόσυρση της οδηγίας για την ε, άδεια μητρότητας. Περιμένουμε νέες νομοθετικές προτάσεις επί του θέματος αυτού από την Κομισιόν. Δεν ξέρω αν τους επόμενους έξι μήνες σκοπεύετε να προβείτε σε συζητήσεις με την ε, Κομισιόν προκειμένου να προχωρήσουν αυτά τα δύο θέματα. Δύο θέματα. Δηλαδή, σας έθεσα το ζήτημα των ε, ε, γυναικών στα διοικητικά συμβούλια και την, ε, της προσωπική προσωπικής και επαγγελματική ζωής. Ευχαριστώ εκ μέρους του EFDD, και Γιούτα. Λοιπόν, ε, και εγώ σας καλωσορίζω εκ μέρους της πολιτικής ομάδας FTD. Ε, απλά και εγώ θα επαναλάβω όλα αυτά τα οποία ελέγχθησαν από τους συναδέλφους. Γιατί ακόμα και αν έχουμε διαφορετικές απόψεις ε, για το περιεχόμενο των προτάσεων, παρόλα αυτά για όλους μας τα επίγοντα θέματα είναι ακριβώς τα ίδια. τώρα λοιπόν βρισκόμαστε και πάλι σε καλές προθέσεις. Ε, σε έξι μήνες ε, είναι αδύνατον να προχωρήσουν σοβαρά τουλάχιστον κάποια θέματα. Αυτό που με πιέζει και θέλω να σας ρωτήσω είναι το εξής. Στο Συμβούλιο ίσως ε, μπορείτε να τους μεταφέρετε και δική μας την άποψη επ' αυτού. Δηλαδή, Όσον αφορά τις πραγματικές ανάγκες των γυναικών, τι ακριβώς πιστεύουν οι κυβερνήσεις. Σας θα σας αναφέρω ένα παράδειγμα. Εχθές, ας πούμε, στην Ιταλία η κυβέρνηση σε σχέση με τη χρηματοδότηση της ημέρας αναπαραγωγής αποφάσισε η κυβέρνηση να δώσει κίνητρα στις γυναίκες για να κάνουν παιδιά μέχρι ή πριν την ηλικία των 30 ετών. Αλλά από ό,τι φαίνεται δεν έχουν καταλάβει γιατί οι γυναίκες τελικά πολύ συχνά δεν μπορούν να κάνουν παιδιά πριν από τα 30. Έχουν πολλές δυσκολίες. Είναι δύσκολο για τις γυναίκες να συμβιβάσουν την ιδιωτική τους με την επαγγελματική τους ζωή είναι δύσκολο να συνδυάσουν τη ζωή ενός μωρού με τη δουλειά τους. Ε, υπάρχουν ε, και θέματα γυναικείας ανεργίας. Άρα δηλαδή, εγώ θέλω να ρωτήσω, τα κράτη-μέλη τελικά τι πιστεύουν, ποια είναι η άποψή τους. Γιατί αν αυτά τα αποτελέσματα μας προσφέρουν, μάλλον μας οδηγούν στην απελπισία. Ίσως εσύ μπορείτε να μεταφέρετε τις ανησυχίες μας στο Συμβούλιο, να τους κάνετε να καταλάβουν ότι κάθε χρόνο λέμε τα ίδια πράγματα. Επαναλαμβάνουμε συνέχεια τα ίδια, γιατί δυστυχώς μέχρι τώρα από ό,τι φαίνεται δεν μπορέσαμε να βρούμε κάποιες λύσεις. Ευχαριστώ πολύ. Τώρα, θα ήθελα να ρωτήσω αν υπάρχουν άλλα μέλη της Επιτροπής που θα ήθελα να λάβουν το λόγο για να θέσουν ερωτήματα. Δεν έχουμε και πολύ χρόνο στη διάθεσή μας. Δύο-τρεις ακόμη ομιλητές. Θα ήθελα να σας ζητήσω να είστε όσο το δυνατόν πιο ε, σύντομοι για να έχει και ο υπουργό χρόνο για να απαντήσει. Κύριε Χάνιμπαλ, ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ κύριε Υπουργέ, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Μιας και αναφερθήκατε στην έκθεση για τις ε, ε γυναίκες στη μετανάστευση, θα ήθελα ε, να σας υπενθυμίσω κάποια πράγματα. Η έκθεση αυτή αποτελούσε τρία, ε, αποτελούνταν από τρία τμήματα. Τη μετανάστευση, την, αυτή καθεαυτή, τα κέντρα υποδοχής και στη συνέχεια η ένταξή τους στην κοινωνία. Ένα από τα ζητήματα που μας απασχόλησαν ήταν η βία κατά των ε, γυναικών σε όλα τα στάδια της μετανάστευσης. Ε, και αυτό που μας ε, απασχόλησε ιδιαίτερα ήταν οι συνθήκες υγιεινής, η ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, η παροχή διερμηνέων για τις γυναίκες πρόσφυγες και μετανάστες και τέλος το ζήτημα των, της κοινωνικής τους ένταξης. Φυσικά το ζήτημα αυτό είναι ευρύτατο και δεν πρόκειται να αντιμετωπιστεί εύκολα και γρήγορα. Θα συνεχίσουμε να έχουμε ε, μεταναστευτικές ροές προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα ήθελα να σας ρωτήσω τι σκοπεύετε εσείς να κάνετε για να αντιμετωπιστούν αυτά τα προβλήματα και ε, τι είδους ε, διάλογο σκοπεύετε να κάνετε στο Συμβούλιο επί αυτών των θεμάτων και θα ήθελα να σας παρακινήσω να συνεχίσετε το διάλογο με τη δική μας Επιτροπή για αυτά τα ζητήματα. Ευχαριστώ Κύριε Μπεσεράνο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Υπουργέ. Έχω μια πολύ συγκεκριμένη πρόταση, ε, ερώτηση. Από τότε που αναλάβατε την ε, Προεδρία του Συμβουλίου, έχετε την αίσθηση ότι υπάρχει βούληση προκειμένου να προχωρήσει ο φάκελος για τις γυναίκες στα διοικητικά συμβούλια. Είναι ένα ζήτημα στο οποίο εμείς ε, έχουμε κατακτήσει ένα πολύ υψηλό επίπεδο συμφωνίας. Είναι ένα ζήτημα που μας απασχολεί και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ε, και εσείς ε, σκοπεύετε να σημειώσετε πρόοδο σε αυτό το θέμα. Ευχαριστώ και τέλος κύριος Σεβάστιαν. Ευχαριστώ κύριε Υπουργέ ομολογώ ότι με ανησύχησαν τα λόγια σας για την κύρωση της Σύμβασης της Κωνσταντινούπολης. Είπατε ότι θα ξεκινήσουν οι διαπραγματεύσεις και έχουμε ακούσει εδώ στην Επιτροπή μας την Επίτροπο Γιουρόβα να λέει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση σκοπεύει φέτος να υπογράψει τη συγκεκριμένη σύμβαση. Υπάρχει μια αντίφαση μεταξύ των όσων μα είπε η Επίτροπο και των όσων μα είπατε εσεί η συγκεκριμένη σύμβαση είναι ένα από τα καλύτερα ε, εργαλεία που έχουμε στα χέρια μας για την κατεπολέμηση της βίας κατά των γυναικών. Ε, είναι σήμερα 1η Σεπτεμβρίου, δεν έχουμε και πολύ χρόνο πια. Θέλω να μου πείτε ακριβώς πού βρισκόμαστε σε σχέση με το συγκεκριμένο θέμα. Ευχαριστώ. Και τώρα ο λόγος στον Υπουργό για να απαντήσει στα ερωτήματα που τέθηκαν. Δέκα λεπτά έχετε κύριε Υπουργέ στη διάθεσή σας. Ευχαριστώ πολύ. Νομίζω λοιπόν ότι μπορούμε να συμφωνήσουμε όλοι μας ότι 10 λεπτά είναι πολύ λίγα. Δεν φτάνουν για να δώσει κανείς ε, επαρκείς απαντήσεις. Ε, ζητώ λοιπόν συγγνώμη ευθύς εξ αρχής ότι δεν θα μπορώ να μπω σε βάθος σε όλες τις ερωτήσεις. Όσον αφορά τώρα τις ερωτήσεις ε, σχετικά με τα δικά μας τα εθνικά, τα σλοβακικά, θα σας στείλω μία επιστολή ε, και μπορώ να σας καλέσω και να συναντηθούμε. Αυτά τα θέματα ευχαρίστως να τα συζητήσουμε ε, κατηδίαν γιατί εκτός από αυτά τα 30 ευρώ ε, θα υπάρξουν και κάποιες άλλες αυξήσεις και όταν μιλάμε για το γεγονός ότι η μητέρα φροντίζει τον άπειρο παιδί της, στην περίπτωση αυτή η μητέρα έχει και δικαίωμα σε σύνταξη ε, ειδική σύνταξη. Ο Υπουργό Οικονομικών το εξτάζει το θέμα και, εν πάση περιπτώσει, ε, και εγώ ευχαρίστω να το συζητήσω μαζί σα. Ε, σα ευχαριστώ πολύ για τι δραστηριότητε που αναπτύσσετε εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ε, και για τι δραστηριότητέ σα στη Σλοβακία. Νομίζω ότι υπάρχει περιτόριο για πάρα πολλά ακόμα που μπορούν να γίνουν πάρα πολλά. Θα ήθελα λοιπόν να ε, ξεκινήσω με θέματα ε, βασικής προσέγγισης. Αναφέρθηκα στο τρίο ε, προεδρίας. Εμείς προτιθέμεθα να αναπτύξουμε δραστηριότητες στο πλαίσιο αυτής της Τρόικα Προεδριών. Μερικές φορές ξεκινάνε ορισμένα πράγματα, αλλά τελικά δεν ολοκληρώνονται. Εμείς ε, Έχουμε επικοινωνήσει σε ανώτατο πολιτικό επίπεδο. Έχουμε έρθει σε επαφή με την Επίτροπο κυρία Τάισεν και μας ε, ενδιαφέρει να προετοιμάσουμε ορισμένα πράγματα έτσι ώστε αν τελικά η Ολλανδική Προεδρία δεν μπορέσει να ολοκληρώσει ορισμένα πράγματα μετά θα ακολουθήσουμε εμείς και ίσως μπορείτε ε, όλα αυτά τα θέματα να τα έχετε κατά νου. Εγώ ε, υπάρχουν πολλά θέματα ε, που θέλω να συζητήσω με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή νομοθετικά και μη νομοθετικά. Κατά τα άλλα, πρέπει να σας πω ότι εκτιμώ ιδιαίτερα αυτά που ανέφερε η Ολλανδική και που έκανε η Ολλανδική Προεδρία. Σημειώθηκε πρόοδος, αλλά υπάρχουν ακόμα θέματα που εκκρεμούν. Και πιστεύω ότι τελικά εμείς ε, θα μπορέσουμε να επιτύχουμε αποτελέσματα μέχρι να ολοκληρωθεί η δική μας η Προεδρία. Όταν μιλάμε για ισότητα των δύο φύλων και για θέματα ποιότητας ζωής, ε, προφανώς ε, μιλάμε για προτεραιότητες ε, που αναφέρθηκαν και χτες στην Επιτροπή Απασχόλησης. Όταν μιλάμε για το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο, για τα κοινωνικά δικαιώματα, αυτό είναι ένα είδος υπέρ δομής, πολύ σημαντική βέβαια, αλλά θέλω να επαναλάβω μία σειρά θεμάτων που ανέφερα εχθές. Υπάρχει λοιπόν μία ολόκληρη σειρά προτεραιοτήτων ε, που αυτές σχετίζονται άμεσα με το γεγονός ότι είμαστε ιδιαίτερα φιλόδοξοι όσον αφορά όλα τα θέματα. Εμείς ε, θέλουμε να κάνουμε πάρα πολλά, ε, θέλουμε να προχωρήσουμε ακόμα περισσότερο, ε, θέλουμε να οργανώσουμε πολλές εξειδικευμένες θεματικές συνεδριάσεις στην Πρατισλάβα. Το θέμα δεν είναι μόνο να συμπεριλαμβάνονται κοινωνικοί εταίροι, αλλά και άλλες σημαντικές κοινωνικές ομάδες, οι οποίες ε, δεν έχουν μόνο την ευκαιρία αλλά και την υποχρέωση να συμμετέχουν. Εμείς θέλουμε να σεβαστούμε τις απόψεις τους, τις ε, προτάσεις τους και όλα αυτά θα εκφραστούν μέσα από νομοθετικές προτάσεις. Και υπάρχει και κάτι άλλο το οποίο θέλω να σας προσφέρω, δηλαδή το πώς ε, οι ευρωπαϊκοί θεσμοί ερμηνεύονται από τους πολίτες μας. Έχουμε καταλήξει ότι δεν είναι πάντα θετική η ερμηνεία από πλευράς ε, πολιτών. Γι' αυτό λοιπόν το λόγο και εμείς αποφασίσαμε να κάνουμε περισσότερα πράγματα. Ε, και για, πάλι για αυτό το λόγο το πρώτο άτυπο ε, Συμβούλιο Κοινωνικών Υποθέσεων στο οποίο αναφέρθηκε η κυρία Ζαμπόρσκα αυτό το πρώτο άτυπο συμβούλιο είχε άμεση σχέση με τις εξελίξεις, με την ψηφιοποίηση, με την πρόοδο της τεχνολογίας και έτσι ε, φτάνουμε σε ε, αλλαγές στην αγορά εργασίας, φτάσαμε σε αλλαγές, κάποια επαγγέλματα εξαφανίστηκαν και νομίζω να σας πω τι έγινε. Εγώ πήγα τους υπουργού σε ένα συγκεκριμένο εργοστάσιο και τους έδειξα τι υπήρχε πριν από 20 χρόνια και τι υπάρχει σήμερα. Κάποια πράγματα εξαφανίστηκαν πλήρως. Είναι λοιπόν πολύ σημαντικό να υπάρχει αυτή η διασύνδεση ανάμεσα στις νομοθετικές προτάσεις και την πραγματικότητα. Και πρέπει να σας πω, με μεγάλη μου χαρά διαπίστωσα ότι όλοι οι υπουργοί που συμμετείχαν σε αυτό το άτυπο ε, συμβούλιο χάρηκαν. Τους άρεσε που πήγαμε σε αυτό το εργοστάσιο. Όσον αφορά τώρα στα συμπεράσματα που έχουν σχέση με τις ε, προτεραιότητες, ο τελικός στόχος είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση να έρθει πιο κοντά στους πολίτες. Έχουμε πετύχει πάρα πολλά αλλά ε, πρέπει να τα πουλήσουμε όλα αυτά με καλό τρόπο στους ε, πολίτες. Ε, και εδώ προσβλέπουμε στη συνεργασία με εσά, θέλουμε να μας βοηθήσετε, να βοηθήσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Αυτά είναι ένα είδος γενικών παρτίσεων και τώρα θα περάσω σε πιο συγκεκριμένες απαντήσεις. Όσον αφορά την συνθήκη της Κωνσταντινούπολης. Μιλάμε για μια μακρά διαδικασία και τώρα πλέον εναπόκειται σε εμά να επιταχύνουμε τη διαδικασία. Εγώ δεν είμαι κατά των προθέσεων της Επιτρόπου να ολοκληρωθεί το όλο θέμα μέχρι το τέλος του έτους, αλλά η δική μας υποχρέωση είναι να προχωρήσουμε τη διαδικασία η οποία δεν βρίσκεται στην αρχή της αλλά έχει ήδη εξελιχθεί. Υπάρχουν κάποια θέματα ε, τα οποία έχουν αναφερθεί. Είπατε και ρωτήσατε κατά πόσον η Ευρωπαϊκή Ένωση θα υπογράψει αυτή την συνθήκη στο σύνολό της. Η απάντηση είναι ναι. Ναι, όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Σλοβακία έχει αποφασίσει να ε, καταρτήσει νόμο που θα αφορά στη βία λόγω της διάστασης και λόγω του διαχωρισμού των δύο φύλων. Εμείς πιστεύουμε ότι είναι πολύ σημαντικό να γίνουν συγκεκριμένα βήματα από το να υπάρξει μόνο αυτή η μακρά διαδικασία κύρωσης. Εμείς θέλουμε κάποια συγκεκριμένα θέματα να τα συμπεριλάβουμε στην εθνική μα νομοθεσία. Και τα χαρώ πάρα πολύ. Αν τελικά σε αυτή την προσπάθεια συμμετέχετε όλοι σας, ε, αυτό βέβαια προποθέτει ε, διεξοδικέ συζητήσει. Μία από τι προτεραιότητές μα είναι να φτάσουμε πιο κοντά στην κύρωση τη σύμβαση. Βεβαίως η σύμβαση θα χρειαστεί περισσότερο χρόνο σε διάφορα εθνικά επίπεδα. Είναι μια μακρά διαδικασία και είναι και μια ατομική, ειδική του καθενός προσέγγιση. Ο στόχος αυτός είναι φιλόδοξος. Ε, ξέρω ότι ορισμένοι από εσά ε, ήδη μπορεί να είσαστε απογοτευμένοι ε, πιστεύετε ότι υπάρχουν ε, ε, κάποια θέματα διακρίσεων που εξακολουθούν να υφίστανται ε, όπως ας πούμε για τη θέση των γυναικών στα εποπτικά και διοικητικά συμβούλια. Συμφωνώ μαζί σας επ' αυτού. Το ίδιο ισχύει και για την οδηγία για την απόσπαση γυναικών. Η Κομισιόν δεν αντιδρά ε, πολλές φορές, κλείνει τα μάτια της, ε, αγνοεί ορισμένα πράγματα και αυτό σημαίνει ότι υπάρχουν θέματα που έχουν συζητηθεί εδώ και 6-7 χρόνια και ορισμένα πράγματα δεν λαμβάνονται υπόψη. 11 ε, κρατημέλη έχουν υψώσει κίτρινη κάρτα ε, σε ένα πολύ σημαντικό θέμα όπως είναι η οδηγία και η οδηγία είναι απαραίτητη για ορισμένα κρατημέλη. Νομίζω λοιπόν ότι δεν, δεν υπάρχει πάντα καλή προετοιμασία πριν ε, ξεκινήσουν νομοθετικές ε, προτάσεις και αυτά ισχύουν και για άλλα θέματα. Αυτά λοιπόν όσον αφορά τις γυναίκες ε, στα εποπτικά διοικητικά συμβούλια. Εμείς τα χαρούμε πάρα πολύ εάν τελικά στο τέλος της προεδρίας μας ε, υπάρξει πρόοδος και αν μπορέσουμε να προχωρήσουμε ακόμα περισσότερο αυτό θα είναι πραγματικό επίτευγμα. Δεν υπάρχει πολλής χρόνος. Να δώσω ποιες ερωτήσεις θα απαντήσω. Είπατε ότι οι γραπτές μας ε, προτεραιότητες ε, φαίνονται καλές, αλλά ότι στην πράξη τα πράγματα δεν είναι τόσο καλά. Ας το δούμε από μια άλλη σκοπιά. Το τρίο προεδριών. Οι Ολλανδοί ξεκίνησαν κάποια, ε, κάποιους φακέλους, τους οποίους εμείς μπορεί να μην τους παραθέτουμε ρητός, αλλά φυσικά και θα συνεχίσουμε το έργο. Το ίδιο ισχύει και για την Επιτροπή Απασχόλησης. Παρέστηκε ο Μαλτέζος Υπουργός και έχουμε ήδη συμφωνήσει για το ποια διαδικασία θα ακολουθηθεί προκειμένου να προχωρήσουν όλοι αυτοί οι φάκελοι. Θέλουμε να, δείτε δηλαδή τη συνολική εικόνα του τρίου προεδριών και αυτό ίσως απαντά και σε ορισμένα από τα δικά σας ερωτήματα. Ίσως γι' αυτό ε, δεν βλέπετε θέματα που θα σας ενδιαφέραν στην, ε, στις προτεραιότητες της Σλοβακικής Προεδρίας. Έξι μήνες είναι πολύ μικρό διάστημα για να ξεκινήσει κανείς μια διαδικασία και να την ολοκληρώσει κιόλα. Αν ε, ιδίω λάβει υπόψη του κανεί και τι πολύ περίπλοκε διαδικασίε που πολλέ φορέ χρειάζεται να, να πραγματοποιήσουμε θεσμικά. Και θα ήθελα να σας ε, υπενθυμίσω ότι τα σεμινάρια, οι συνεδριάσεις και οι εκδηλώσεις που θα γίνουν στην Πρατισλάβα είναι πολύ σημαντικά και θα ήθελα για άλλη μια φορά να επαναλάβω την πρόσκλησή μου προς εσάς για να παρευρεθείτε στις εκδηλώσεις αυτές. Ευχαριστώ πολύ κύριε Υπουργέ για τις απαντήσεις σας και σας ευχαριστώ και για την πρόσκληση που μας απευθύνατε να συμμετάσχουμε στις εκδηλώσεις αυτές. Εμείς τώρα θα συνεχίσουμε, θα κάνουμε ένα πεντάλεπτο διάλειμμα για, ε, και στη συνέχεια θα συνεχίσουμε με την ημερησία διάταξη μας.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 Vážené kolegyne, kolegovia, poprosila by Συνάδελφοι, σας παρακαλώ καθίστε. Θέλω να συνεχίσουμε με την ημερήσια διάταξη. Οι διερμηνείς μας παραχώρησαν άλλα 15 λεπτά. Μετά τις 11 αλλά οι συντονιστές συνεδριάζουν κανονικά στις 11, οπότε παρακαλώ να είστε συντομότατοι. Κύριε Μπεθέρα, η συγγήτρια έχει το λόγο. Ναι, θα είμαι πάρα πολύ σύντομη. Γιατί 1η Σεπτεμβρίου έχουμε και θα πρέπει να προχωρήσουμε και με άλλα ζητήματα με τους συντονιστές. Έχουμε το σχέδιο, δεν έχουμε ακούσει το σκιώδη, τους σκιώδης εισηγητές ακόμη ποια άποψη έχουν. Θα ήθελα λοιπόν να σκεγγραφίσω λίγο το περιεχόμενο της έκθεσης και να επανέλθω στους στόχους. Ε, νομίζω ότι έτσι μπορούμε να επιτύχουμε καλύτερα αποτελέσματα αν έχουμε μια πληρέστερη εικόνα. Ευχαριστώ τους εισηγητές από τις διάφορες πολιτικές ομάδες ε, που έλαβαν το σχέδιο της έκθεσής μου πριν από τις καλοκαιρινές διακοπές. Με το που συλλέξω τις απόψεις ε, των εισηγητών ε, θα στείλω το κείμενο στη μετάφραση και τον Οκτώβριο θα σας παρουσιάσω το ολοκληρωμένο κείμενο και μετά μέχρι τον Νοέμβριο θα καταθέσετε εσείς τις τροπολογίες σας. Τέλη Νοεμβρίου θα γίνει ψηφοφορία και το Δεκέμβριο θα περάσει την Ολομέλεια. Αυτό είναι το χρονοδιάγραμμα. Επιτρέψτε μου τώρα να επανέλθω στην γενική προσέγγιση που υιοθέτησα για την έκθεσή μου προώθηση τη ισότητα των Φίλων για το θέμα των κλινικών δοκιμών και της ψυχικής υγείας. Αυτός είναι ο τίτλος. Βασόμαστε στην ορισμό του ΠΟΕ για την ψυχική υγεία Ε, και δεν μιλάμε μόνο για απουσία ασθενειών ε, ή νοσημάτων, αλλά για ένα εύση είναι μια κατάσταση καλής υγείας. Ε, έχουμε προβλήματα ως προς την πρόσβαση στις πληροφορίες, στην πρόσβαση στις υπηρεσίες του τομέα υγείας. Οι γυναίκες έχουν δε ιδιαίτερες ανάγκες για την σεξουαλική και αναπαραγωγική τους υγεία. Η έρευνα και οι πρακτικές δεν λαμβάνουν όντως υπόψη τις διαφορές ε, ανάμεσα στους, στις γυναίκες και τους άντρες ως προς ε, το είδος ε, των υπηρεσιών που χρειάζονται μεν και η δε. Το 50% λοιπόν του ευρωπαϊκού πληθυσμού υποεκπροσωπείται στη ιατρική έρευνα. Οι έρευνες παίρνουν σε δεδομένο την τέλεια ισότητα των δύο φύλων δεν λαμβάνουν υπόψη όμως τον, τους κοινωνικούς παράγοντες που επηρεάζουν ε, την υγεία. Οι θεραπευτικές αγωγές ε, των ε, γυναικών έχουν δοκιμαστεί σε άντρες και αυτό δεν είναι αποτελεσματικό, μπορεί δεν να αποβεί και αντιπαραγωγικό. Χρειαζόμαστε λοιπόν κονδύλια για την έρευνα που προέρχονται από τον κρατικό προϋπολογισμό από τα χρήματα των φορολογουμένων. Για την ψυχική υγεία έχουμε δεδομένα από ψυχιατρικές κλινικές, είναι συγκρίσιμα τα δεδομένα για τα δύο φύλλα, όμως η τυπολογία των νοσημάτων ε, είναι εντελώ διαφορετική. Το άγχος και η κατάθλιψη είναι πολύ συχνότερο φαινόμενο στις γυναίκες ε, στην υγειονομική πολιτική, στην πολιτική στον τομέα Υγεία των κρατών μελών δεν λαμβάνονται υπόψη, όντως ξαναλέω, οι διαφορές των δύο φύλων. Τι είναι οι βασικοί άξονες της έκθεσής μου και θα ήθελα όλοι να προβληματιστούμε για αυτά τα ζητήματα. Το θέμα τη υγεία ενσωματώνει σε όλες οι υπόλοιπε πολιτικές Ευρωπαϊκή Ένωση, για την πρόληψη των ασθενειών, για τον περιορισμό των πηγών κινδύνου, για την υγεία, είτε πρόκειται για σωματική είτε για ψυχική υγεία. Όλοι θα πρέπει να υπομισθούμε αυτή την ευθύνη η καθολική πρόσβαση σε ποιοτικέ υπηρεσίες και η αλληλεγγύη είναι επίσης σε κοινέ αξίες ε, των οποίων θα πρέπει να εδράζεται το σύστημα υγείας των κρατών μελών. Η ισότητα των φύλων συνεπάγεται και η ισότητα πρόσβασης στις υπηρεσίες ανεξαρτήτως εθνοτικής προέλευσης, ε, ηλικίας, ε, κοινωνικής τάξης, ε, οικονομικών μέσων. Εξάλλου το εγγυάται η χάρτα των θεμελιωδών δικαιωμάτων, εγγυάται καθολική πρόσβαση στις ιατρικές επί τη βάση των συνθήκων ε, που ισχύουν σε κάθε κράτος μέλος και των εθνικών πρακτικών. Φυσικά θα πρέπει να ληφθούν υπόψη ε, τα όσα προβλέπονται ε, και διαφορά για την ισότητα των δύο φύλων στις συμβάσεις σε συνθήκες Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ξαναλέω, θα πρέπει σε τις πολιτικές να ληφθούν υπόψη τα ιδιάζοντα χαρακτηριστικά των δύο φύλων για να εκπονηθούν σωστά οι πολιτικές στον τομέα της υγείας. Κλείνοντας, θα ήθελα να υπενθυμίσω πως ε, η Γενική Κατεύθυνση ε, από πλευρά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, είναι να ληφθεί απόψη, ε, υπόψη, να ληφθούν υπόψη οι πληροφορίες που προκύπτουν από διάφορες μελέτες που έχουν γίνει. Όμως στην πράξη προς το παρόν δεν έχουν γίνει πρακτικές ρυθμίσεις για να ικανοποιήσουμε τις ανάγκες του μισού πληθυσμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εξακολουθούν αυτοί που εκπονούν τις πολιτικές να αγνοούν την διάσταση αυτή. Ε, αυτό αντιβαίνει πλήρω στι συνθήκε λειτουργία Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτά εν γέννη, ανέκει και για την δομή τη έκθεση, θα το είδατε στο έγγραφο εργασία. Στο μέτρο που θέλουμε να καλύψουμε διάφορα ζητήματα, θα μιλήσουμε και για τα γενικά προβλήματα στον τομέα της υγείας το θέμα της ανισότητας των δύο φύλων, αλλά θα έχουμε και ένα συγκεκριμένο τμήμα ειδικού ε, για, το, για την ψυχική υγεία και ένα τρίτο τμήμα είναι πάρα πολύ σημαντικό κατά την άποψή μου. Ένα τρίτο τμήμα, διότι συνδέεται με διάφορε θεματικέ ενότητες που μας ενδιαφέρουν, ναι, μεταξύ των οποίων το πιο σημαντικό είναι οι κλινικές δοκιμές και η χρήση των ευρωπαϊκών κονδυλίων για την διεξαγωγή αυτών των δοκιμών, ε, συνθήκες πλήρης διαφάνειας. Ιδού, θα σταματήσω εδώ. στη διάθεσή σας για ερωτήσεις οι σκιώδεις θα έχουν τη δυνατότητα να μου διαβάσουν τις απόψεις τους ε, για να βελτιώσω το σχέδιο έκθεσης. Ελπίζω σύντομα να γίνει σύσκεψη των σκιωδών για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε. Ευχαριστώ πολύ για την έκθεσή σας αυτή και για την παρουσίαση. Τώρα θα ήθελα να δώσω το λόγο στους ε, σκιώδεις των πολιτικών ομάδων. Δεν υπάρχει κανείς από το ΕΛΚ εδώ, οπότε μπορούμε να ξεκινήσουμε με τους σοσιαλιστές. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ. Έχω διαβάσει όλα τα έγγραφα, συγγνώμη διατρες που ήρθα λίγο αργά. Με έχεις εντυπωσιάσει. Θέλω να σας ευχαριστήσω για το έγγραφο εργασίας, ιδίως γιατί νομίζω ότι θα διευκολύνει το έργο μας. Και χαίρομαι πολύ που συμμετέχω σε αυτήν την ε, ομάδα, γιατί έχω ασχοληθεί μέσω πολιτιστικών ε, δραστηριοτήτων, μέσω του θεάτρου και των τεχνών με ζητήματα ψυχικής υγείας, με ανθρώπους που αντιμετωπίζουν προβλήματα ψυχικής υγείας και εγώ στην ε, χώρα μου έχω ξεκινήσει και το φόρουμ για την ψυχική υγεία και το να εξετάσουμε αυτό το θέμα και από την σκοπιά του φίλου είναι πολύ σημαντικό. Υπάρχουν ε, ζητήματα φίλου στο ευρύτερο θέμα της, της ψυχικής υγείας και χρειαζόμαστε μια ολιστική προσέγγιση, ε, μια προσέγγιση που θα εξετάζει ολόκληρη την κοινωνία και αυτό συνάδει και με τη στρατηγική του ΠΟΗ για το διάστημα 2017-2021. Πολλοί συνάδελφοι έχουν πει ότι ζητήματα όπως το άγχος, η κατάθλιψη, ε, ο πανικός, ε, η κρίση πανικού ε, πολλές φορές πλήττουν σε μεγαλύτερο βαθμό τις γυναίκες από τους άντρες γιατί ακριβώς αποτελούν ένα, ένα ζήτημα που μπορεί να θέσει σε κίνδυνο και την ευμερία των γυναικών. Ε, είναι ανάγκη λοιπόν να αντιμετωπιστούν και αυτά τα θέματα. Η ψυχική υγεία εξακολουθεί να είναι ένα ζήτημα που χαρακτηρίζεται από ένα κοινωνικό στίγμα. Μόνο ε, ε, δύο από τους, μόνο το 20% όσων αντιμετωπίζουν προβλήματα ψυχικής υγείας ζητούν βοήθεια. Πολλές φορές γυναίκες και κορίτσια προσπαθούν να τα αντιμετωπίσουν μόνες τους αυτά τα προβλήματα και αυτό επιτείνει ε, την οξύτητα των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν. Πολλές φορές γυναίκες οι οποίες ε, ε, Ιδίω αυτό αφορά και τις γυναίκες στην τρίτη ηλικία, ιδίω όταν χάνουν τους συντρόφους τους. Χρειάζεται να ενισχύσουμε την ευαισθητοποίηση και να συνδέσουμε τις πολιτικές για την ψυχική υγεία και για την, για την ισότητα των ε, ε φύλων. Ε, η, ε, ο πολυδιάστατος χαρακτήρας του κοινωνικού αποκλεισμού και της ισότητας των φίλων ε, μας οδηγεί στο ότι πρέπει να εξασφαλιστεί η πρόσβαση σε υπηρεσίες ψυχικής υγείας ιδίως στο επίπεδο των δήμων και των κοινοτήτων, μορφές παρέμβασης που θα πρέπει να δημιουργηθούν, υποστηρικτικές που ε, στο Ηνωμένο Βασίλειο ε, χρησιμοποιούμε και τον όρο της ε, κοινωνικής συνταγογράφησης, όπου μπορεί ένας γιατρός δηλαδή να παροτρύνει έναν ασθενή ε, να ασχοληθεί με δημιουργικές ε, εργασίες όπως είναι η συγγραφή για παράδειγμα. Όλα αυτά βεβαίως ε, έχουν και ένα κόστος και εν πάση περιπτώσει εγώ θα ήθελα να σας πω ότι χαίρομαι πολύ που θα συνεργαστούμε στο θέμα αυτό. Ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Μπιόρκ έχει το λόγο. Thank you. Θα είμαι πάρα πολύ σύντομη. Το διάβασα και εγώ το σχέδιο έκθεσης ε, και προσβλέπω μια ανυπομονησία στη συνεργασία μας για αυτή την έκθεση. Θεωρώ είναι πολύ καλή η δομή και μπορούμε να βασιστούμε σε αυτή για τις μελλοντικέ ε, εργασίες. Ε, ενδεχομένως, δεν ξέρω πόσο χρόνο θα έχουμε, θα ήθελα να μιλήσουμε και για το θέμα του burnout, πολύ συχνό φαινόμενο στη Σουηδία και όχι μόνο. Ε, είναι η επαγγελματική ζωή των γυναικών ε, ε, φορτωμένη σε σχέση με την οικογενειακή του ζωή και Βλέπουμε επίσης ότι οι γυναίκες που δουλεύουν σε τέτοιες κλινικές και σε Ε, ε, υποφέρουν οι ίδιες από εξάντληση και ε, από προβλήματα ψυχικής υγείας. Θα ήθελα και αυτό, αν μπορείτε να το συμπεριλάβετε. Ευχαριστώ, κύριο Σεμπάστιν. Ευχαριστώ πολύ. Και εγώ μιλώ εξ ονόματος της Επιτροπής Ανάπτυξης η οποία χαίρεται πάρα πολύ για το ότι έχουμε ή μπορούμε να ε, τοποθετηθούμε πάνω σε αυτή την έκθεση με γνωμοδότηση. Εχθές ε, παρουσίασα εγώ την άποψή μου στην Επιτροπή μου. Οι αντιδράσεις ήταν πολύ θετικές και πρόκειται για το εξής. Μας ενδιαφέρει να συγκεντρώσουμε όλες τις ε, απόψεις. Ε, υπάρχουν βέβαια δύο θέματα τα οποία μας ενδιαφέρουν ιδιαίτερα. Υπάρχει αυτή η διασύνδεση ανάμεσα στη φτώχεια και τις γυναίκες, ότι οι γυναίκες είναι πιο φτωχές από τους άνδρες και αυτό λοιπόν σημαίνει ότι υπάρχουν κάποιες ασθένειες που παραμελούν και που αφορούν κυρίως τις γυναίκες. Πράγματι υπάρχουν ευρωπαϊκές πολιτικές που αφορούν στην έρευνα αυτών των ασθενειών, όμως τα αποτελέσματα της έρευνας δεν διατίθενται. Νομίζω ότι η πολιτική πολιτική ε, υγείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να αναθεωρηθεί. Εμείς θα καταθέσουμε ε, σχετική τροπολογία. Και να πω και κάτι άλλο. Ε, σε μεγάλο βαθμό είμαστε υπεύθυνοι για το θέμα της μετατόπισης ιατρικών δοκιμών στην Αφρική. Επ' αυτού υπάρχουν πάρα πολλά έγγραφα, υπάρχουν και πολλές σχετικές ταινίες ιατρικές ε, λοιπόν προσπάθειες ε, ε, οι οποίες μεταφέρονται όλες στην Αφρική και ο λόγος είναι πάρα πολύ σαφής ότι στις χώρες αυτές παραβιάζονται άνετα τα δικαιώματα των ανθρώπων. Πάρα πολλές λοιπόν γυναίκες στην Αφρική γίνονται ε, ινδικά χειρίδια, ένα είδος πειραματόζων. Χαίρομαι πάρα πολύ για όλη αυτή την πολύ καλή δουλειά και η Επιτροπή Ανάπτυξης χαίρεται πάρα πολύ ε, που συμμετέχουμε και εμείς στην εκπόνηση της έκθεσης. Αυτό μας ε, μοιάζει πάρα πολύ σημαντικό. Ευχαριστούμε πολύ. Δυστυχώς δεν έχουμε πάρα πολύ χρόνο στη διάθεσή μας, αλλά παρόλα αυτά ε, θα ήθελα να δώσω το λόγο στην ε, εισηγήτρια. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ ε, για τις παρεμβάσεις των συναδέλφων. Ευχαριστώ και για αυτά που είπαν οι συνάδελφοι της Επιτροπής Γενικών και από την Επιτροπή Ανάπτυξης. Νομίζω ότι αυτό που ενδιαφέρει κυρίως είναι το θέμα των πειραμάτων για τα φάρμακα. Ε, ε για αυτό το θέμα. Ε, πολύ ασχολούμεθα με το θέμα αυτό, άρα δηλαδή αυτό σίγουρα θα το συμπεριλάβουμε στις εργασίες μας. Και θα δούμε μήπως ε, μπορούμε όλοι από κοινού να συνεργαστούμε για να δούμε τι θα κάνουμε και μετά θα προχωρήσουμε.